Uh, Κυρίες και κύριοι, είναι ήδη μισή, οπότε θα ξεκινήσουμε σχεδόν αμέσως. Καθίστε παρακαλώ. Έχουμε το επιτελείο των περισσότερων εισηγητών και σκιωδών εισηγητών μας. Κυρία Γκέπχαρτ, θα έρθει ο κύριος Πέρες, ε, Πέρες, ή θα αντικαταστήσετε εσείς σκιώδη συγγετρία. Για να ξεκινήσουμε με την έκθεση του κυρίου Διόν. Right. Um, well, good morning everybody. Um... Ωραία, καλημέρα σας. Θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της πρώτης μέρας από τη διήμερη συνεδρίασή μας, καλωσορίζοντας ε, τα μέλη της Επιτροπής και φυσικά και όσοι μας παρακολουθούν ε, από το διαδίκτυο. Κάποιες ε, ανακοινώσεις πρώτα. Καταρχήν έχετε λάβει το νέο newsletter θα το βρείτε και στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να το λαμβάνετε και στο κινητό σας. Είναι πηγή πολύ χρήσιμα πληροφοριών. Επίσης, έχουμε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους ε, της Διεύθυνσης Επικοινωνιών για να βελτιώσουμε την πρόσβαση των συναδέλφων στα έγγραφα, γιατί τίνουμε προς μία συνεδρίαση χωρίς ε, έγγραφα για λόγους οικονομίας. Επίσης, είμαστε και στο μήνα της εσωτερικής αγοράς για το 2013 που επίσημα ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου. Οπότε, αν πάτε στο yourideasforeurope.eu θα δείτε την ε, διαδικτυακή ανταλλαγή απόψεων που γίνεται με προτάσεις για τη βελτίωση της ε, εσωτερικής αγοράς. Επίσης μπορείτε να συμμετέχετε και σε ε, chat στο διαδίκτυο και μπορείτε να απαντάτε και ζωντανά σε ερωτήσεις των πολιτών. Πολλοί συνάδελφοι το επιχείρησαν χθες και θα ήθελα να πω και στους συντονιστές και στα μέλη ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε τέτοιο chat, μία ώρα είναι η διάρκεια, σας παρατρύνω ένθερμα να το δηλώσετε, γιατί είναι πολλοί που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις για τα δικαιώματά τους ό,τι φορά την εστερική αγορά. Οπότε, αν δεν είχατε αυτήν την εμπειρία, σας παρατρύνω θερμά να το επιχειρήσετε. Και καλωσορίζω και πάλι το κοινό από το διαδίκτυο. Τώρα, ε, καλωσορίζω την Σουζάνα Ρόιτοβα που έχει ασχοληθεί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και έχει επιτελέσει πολύ ε, σημαντικό έργο για πολλά τεχνικά θέματα. Έχω δύο ανακοινώσεις. Καταρχήν, Έχουμε ένα επιπλέον μέτρο για τον εξοπλισμό σε ό,τι αφορά την πίεση. Ίδια αντιμετώπιση θα έχουμε και εδώ. Και οι συντονιστές συμφώνησαν να συμπεριληφθεί και αυτό ε, στο πακέτο που έχει αναλάβει η κυρία Ρόιτοβα. Επίσης, όσοι παρακολουθούν το έργο γνωρίζουν της Επιτροπής, γνωρίζουν ότι είχαμε πρόβλημα στην τελική συμφωνία με το Συμβούλιο για την ε, διατύπωση που προσθέσαμε σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ε, διαδικασίες ε, τροπολογίας και εφαρμογή. Η Λιθωνική Προεδρία με ενημέρωσε για τη νέα συμβαστική πρόταση που βρίσκεται επιτάπητος και που μας ικανοποιεί και ευελπιστούμε ότι θα συμφωνηθεί και στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων τρεχούσης εβδομάδα. Να δώσω όμω καλύτερα πρώτα το λόγο στην κυρία Ρόιτοβα που θα μας ενημερώσει για το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αν φυσικά επιθυμεί η κυρία Ρόιτοβα να λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω νέα, γιατί συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, οπότε δεν έχουμε εξέλιξη. Κυρίως ο βοηθός μου παρακολουθεί το θέμα αυτό και ελπίζω μέχρι την επόμενη εβδομάδα να ολοκληρωθεί το θέμα. Ε, αυτή τη εβδομάδα δεν ήταν εδώ βοηθός γιατί είχε μία γαστρεντερίτιδα. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να μπορέσει να συνεχίσει. Έγινε μία αναβολή της ε, εφαρμογής ε, του όλου πακέτου, κάτι που με δυσαρέστησε λόγω της τελευταίας προσθήκης και της έλλειψης συμφωνίας. Θα ήθελα να σου ζητήσω αν γίνεται να μεταφραστεί αυτό το ενημερωτικό φυλάδιο για τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί μερικές φορές έχουν πρόβλημα και δεν καταλαβαίνουν τι εστί η εσωτερική αγορά. Θα προσπαθήσουμε, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε τους απαραίτητους πόρους. Θα πρέπει να το θέσουμε στην ε, μονάδα ε, επικοινωνιών. Ίσως μία επιτομή να μεταφράζεται. Όχι τις πλήρες εκθέσεις, αλλά τουλάχιστον μια σύνοψη του κοινοβουλευτικού έργου, γιατί συμφωνώ μαζί σου ότι χρειαζόμαστε βελτίωση της επικοινωνίας, όχι μόνο με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά και με τους ενδιαφερομένους γενικώ και την κοινωνία των πολιτών. Και συμμερίζομαι τη δυσαρέσκειά σου για το νέο νομοθετικό πλαίσιο και το έθεσα και στους ε, πρέσβεις των χωρών. Ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε λογικές λύσεις. Τώρα, πριν περάσουμε στο πρώτο θέμα, να σας ενημερώσω για τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου. Τα έχετε λάβει. Αν μέχρι το τέλος συνεδρίας δεν υποβληθούν παρατηρήσεις, θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Έγινε ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους ε, με το προηγούμενο θέμα, γιατί οι μόνες διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται είναι αυτές της κυρίας Ρόιτοβα. Οπότε θα περάσουμε τώρα στην έκθεση της πρωτοβουλίας του κυρίου Κορνέλης Διόγκ, τον καλωσορίζω, για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Λιανικής. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, 90 και κάτι από ό,τι ξέρω, κάτι που δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον που προκάλεσε αυτό το θέμα. Θα δώσω στον εισηγητή το λόγο να σχολιάσει τι τροπολογίε και τι συμβαστικέ προτάσει Να καλωσορίσω την κυρία Ρίβεν και την ομάδα τη από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερική αγορά που παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το δικό μα έργο. Και επίση να σα ε, υπενθυμίσω ότι αύριο το απόγευμα θα έχουμε στην Επιτροπή μα με αναμετάδοση από το διαδικτύο απευθεία την πρώτη στρογγυλή τράπεζα για το λιανικό εμπόριο που σχετίζεται άμεσα με την έκθεση αυτή και θα έχουμε εκπροσώπους ε, και από τον τομέα του λιανικού εμπορίου και από τον τομέα φουδιασμού ε, και σας ε, προσκαλώ στην αυριανή στρογγυλή τράπεζα. Από τους και ηγητές έχουμε τον κύριο Σβάμπ. Θα έρθει σε λίγο και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Η κυρία Πέρες δεν έχει έρθει. Λόκαγκαρτα καθυστέρησε. Η κυρία Ρούλερ όμως είναι παρούσα. Και εγώ είμαι εδώ φυσικά, οπότε έχουμε κρίσιμη μάζα για τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στη συνέχεια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα όμως τον κύριο Ντεγιόμ για να σχολιάσει τις τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ε, κατέθεσαν ε, τροπολογίες. Ε, σίγουρα είμαι σε θέση να εγκρίνω πολλές από αυτές ως ε, ευπρόσδεκτες ε, προσθήκες και βελτιώσεις στο κείμενο. Αναφέρθηκε και στον πρώτο γύρο συζήτησης ότι πολλά μένουν ακόμα να εποθούν για το λιανικό εμπόριο. Πολλές τροπολογίες λοιπόν δεν μου δημιουργούν εμένα τουλάχιστον πρόβλημα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που θα ήθελα να αναφέρω. Βεβαίω ε, θα καταρτήσω και συμβιβαστικέ τροπολογίε στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα, γιατί υπάρχουν και κάποιε επικαλύψει. Σε αρκετέ τροπολογίε. Τώρα, τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, που και πολύ σημαντικό για μένα, είναι οι παράγραφοι που μιλούν για το, το ανεξάρτητο λιανικό εμπόριο, τα μικρά καταστήματα τα είπαμε και την πρώτη φορά που συζητήσαμε την έκθεση. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, τροπολογίες που νομίζω ότι φτάνουν στα όρια. Ε, στην ανησυχία τους κατά του προστατευτισμού. Και την προηγούμενη φορά εγώ δήλωσα ότι δεν είμαι υπέρ του προστατευτισμού, όμως αν εξετάσουμε την πολιτική της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις, έχουμε την απόφαση de minimis της Επιτροπής, που λέει ότι τα κράτη μπορούν να δίνουν ενισχύσεις ε, μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό και αυτό είναι απολύτως νόμιμο. Δεν χρειάζεται να είμαστε ακόμα πιο περιοριστικοί από η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέτρα στήριξης, γιατί αυτό είναι μια κοινή πρακτική δεν χρειάζεται κάθε φορά να μπούμε στη δικασία υποβολής εκθέσεων για αυτή την στήριξη μικρής κλίμακας που είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τους ε, μικρούς λιανεμπόρους και βεβαίως δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις, ούτε να αντιβαίνει στις αρχές ε, του δίκαιου ανταγωνισμού ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό εδώ λοιπόν. Αφενός να πληρούνται όλοι οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων του θεμητού ανταγωνισμού, από την άλλη όμως ε, να μην δυσκολεύουμε και δυσχεραίνουμε και τις τοπικές αρχές ε, να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το τομέα και να στερίζουν το λιανικό εμπόριο. Αυτό είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω. Δεύτερον, πιο οριζόντιο θέμα, πολύ συχνά όταν υπάρχει ε, πρόβλημα στρεφόμαστε προς την Επιτροπή για να το λύσει. Για παράδειγμα, για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν νομίζω ότι είναι καθήκον της Επιτροπής να βοηθήσει κάθε επιχειρηματία να αναπτύξει ένα δίκτυο ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχουμε ολόκληρα δίκτυα επιχειρήσεων, εθνικών φορέων που μπορούν να μας βοηθήσουν. Δεν χρειάζεται να στρεφόμαστε πάντα προς ε, αυτό το κεντροποιημένο πρότυπο. Πολλά κρατημέλη ζητούν από την Επιτροπή να κάνουν δραστηριότητες ε, μικρής κλίμακας στα ίδια τα κρατημέλη. Δεν είναι αυτό το καθήκον της Επιτροπής. Η Επιτροπή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να συγκεντρώνει βέλτες στις πρακτικές, να ανταλλάσσει πληροφορίες, ε, ίσως ε, να βρίσκει κάποια πρότυπα, εργαλεία, αλλά δεν πρέπει να ζητάμε κατά πάντα από την Επιτροπή. Και τέλος, Τελευταία παρατήρηση αφορά μια κατάσταση που έχουμε τώρα και στις κάτω χώρες. Ε, βλέπουμε ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν μπει σε, έναν πόλεμο τιμών ε, που βεβαίως ε, χαροποιεί ιδιαίτερα τους καταναλωτές, ιδίω εν μέσω κρίσης, όμως την ίδια στιγμή μία από τις αλυσίδες υπεραγορών έχει στείλει επιστολή προς τους προμηθευτές δηλώνοντάς του ότι πρέπει να μειώσουν τις τιμέ τους κατά 10-15%. Δεν ξέρω πώ θα το κάνετε, γιατί εγώ ω σούπερ μάρκετ έχω μπει σε ένα πόλεμο τιμών. Αυτό βεβαίω και αντιβαίνει ε, πλήρω ε, στι αρχέ τη ε, εθελούσεω πρωτοβουλία, γιατί πρόκειται για φυστάμενε συμβάσει που ξαφνικά έχουν σπάσει, γιατί τα σούπερ μάρκετ αποφάσισαν να κάνουν έναν πόλεμο αγορών τιμών μεταξύ του. Και αυτό βεβαίω δεν είναι σωστό αμέσως ε, μετά την έναρξη αυτής ε, της πρωτοβουλίας υπάρχει ένα ε, πρόβλημα εάν στο πλαίσιο της εθελοντικής πρωτοβουλίας εξετάσουμε αυτό το θέμα θα μπορούσα να πω ότι θα πρέπει να τη στηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή την πρωτοβουλία, γιατί είναι αποτελεσματική. Αν όμως η πρωτοβουλία αυτή δεν κάνει κάτι ως προς αυτό, αδρανήσει δηλαδή και, εγώ έχω κάνει κάποιες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά τη δράση της πρωτοβουλίας, τότε ε, θα τίνω να καταλήξω σε μια συμβαστική ε, πρόταση που θα ζητά περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις. Γιατί έχω δει τροπολογίες συναδέλφων που ζητούν ε, ρύθμιση της επιβολής. Επίσης, μια άλλη ε, ενδιαφέρουσα ιδέα για τον Ευρωπαϊκό Δημοσιολαβητή. Δεν τα έχω εντάξει αυτά, γιατί εγώ πραγματικά στηρίζω και πιστεύω την ε, πρωτοβουλία. Όμως ε, θα πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά εφαρμόζονται. αν η πρωτοβουλία αποδειχθεί αποτελεσματική αυτή και την επόμενη εβδομάδα, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Γιατί πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση, σχεδόν κρίση θα την αποκαλούσα αυτό που διαδραματίζεται τώρα στις κατοχώρες. Αυτά θα δούμε τι έχουν να πούν και οι συνάδελφοι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας. Διατρέχω τις τροπολογίες και νομίζω ότι πραγματικά ε, υπάρχουν πολλά σωστά σημεία όπως αναφέρατε κι εσείς. Γιατί ξέρουμε ότι με τις ε, ε, εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας υπάρχει και ένας περιορισμός στο κείμενο να δώσουμε το λόγο τώρα στους σκιώδεις. Κύριε Σφάπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Η Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ θα ήθελε να σημειώσει ως και ως εισηγήτρια ότι ήταν πολύ ευχάριστη συνεργασία με τον εισηγητή και θεωρεί πως έχει επιλέξει σωστό δρόμο για την έκθεση αυτή. Είναι ε, επαρκής εν γέννη η έκθεση. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ σε ένα σημείο επισημαίνει ε, έλλειψη στην έκθεση ως προς εμπόδια που εντοπίζονται στην διασυνοριακή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τώρα στη δυνατότητα για ελεύθερη εγκατάσταση και θα ήθελε στο σημείο αυτό να δώσει περισσότερη έμφαση και να μιλήσει για επιπλέον δοκιμές ή για μια αναγνώριση ε, πιστοποιητικών ελέγχου από τις αρχές άλλου κράτους. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να καταγραφούν αυτά, ότι σε διασυνοριακό εμπόριο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Βλέπω ότι και η κυρία Γκέπχαρτ ενδιαφέρεται για θέματα ε, των υπηρεσιών και διαβάζει τις τροπολογίες μας. Νομίζουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους διαφορές στην παροχή των υπηρεσιών σε μια τέτοια εσωτερική αγορά. Επίσης, ρητά αναφέρει η κυρία Κοράτσα Μπίλτ ότι ανεξάρτητος του ποια είναι η δομή του εμπόριου, δηλαδή είτε πρόκειται για ηλεκτρονικό εμπόριο ή είτε πρόκειται για αγορά από κατάστημα, έχουμε να κάνουμε με ανταγωνιστικότητα, αυτό είναι το κύριο δηλαδή ζητούμενο, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την επικράτηση προστατευτικών ε, επιλογών. Ξέρω όμως ότι ο κύριος Ντε Ιόγκ προς την κατεύθυνση αυτή τίνει και τον υποστηρίζουμε. Τρίτον, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα πολύ σημαντικό θεμέλιο στην Ευρώπη. Θέλουμε να το αναπτύξουμε, θέλουμε να του επιτρέψουμε, επιλύοντας τα προβλήματα, να υπηρετήσει την προμήθεια προϊόντων, την παροχή των προϊόντων. Χρειάζεται λοιπόν μία προσεκτική εξέταση και του θέματος των φαρμακευτικών προϊόντων που δεν μπορούν να περνάνε μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Νομίζουμε ότι και αυτό αναφέρεται ε, επαρκώς στην έκθεση. Στην πρώτη εκθέση θέλουμε μια διαφανή ε, δυνατότητα επιλογής για τον καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην τροπολογία όπου γίνεται λόγος για, την, για το ιδιωτικό σήμα η ιδιωτική σήμανση καλύτερα προϊόντων. Θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ε, προστασία του καταναλωτή. Δηλαδή όταν υπάρχει αυτή η ιδιωτική σήμανση να μην επιβάλλεται άνωθεν αλλά να λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή. Στο B2B, business to business, ε, επίσης θέλουμε να κάνουμε τις ίδιες παρατηρήσεις και η κυρία Κοράτσα Μπίρτ μα λέει ότι για την αυριανή εκδήλωση, αύριο το απόγευμα που αναφέρατε και εσεί κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη συμμετοχή σε αυτή την ε, retail round table, στρογγυλή τράπεζα για το λιανεμπόριο, που δυστυχώ δεν μα έχει μεταφραστεί στα γερμανικά. Και ε, με αυτά ολοκληρώνει τι παρατηρήσει τη κυρία Κοράτσα Μπίρτ. Καλώ λέει Η κυρία Πέρες δεν είναι εδώ. Κυρία... Α, ο, ναι, εσύ Ευλίν. Εκ μέρους της ομάδας μου θα ήθελα να σημειώσω ότι ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ντεγιόγκ. Είναι πολύ καλή βάση συζήτησης αυτή η πρόταση. Έχουμε πολύ υλικό και προτάσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Σε ένα θα ήθελα να επιμείνω, δύο μάλλον σημεία. στις τροπολογίες που μας έχουν υποβληθεί και αν θα έχει την καλοσύνη και ο συνάδελφος να με ακούσει, αχ τι καλώς πες, ευχαριστώ, η οδηγία για την παροχή των υπηρεσιών δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί για πράγματα τα οποία δεν προβλέπει η ίδια. Δεν είναι μία οδηγία που προβλέπει ιδιωτικοποίηση, απελευθέρωση, ούτε απαγορεύει κανόνας. Σε αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε το λιανεμπόριο. Δεν θέλουμε να μεταφέρουμε στον τομέα των, ε, του λιανεμπορίου κάτι που δεν προβλέπεται γι' αυτό, δεν είναι ειδικά σχεδιασμένο γι' αυτό. Και επίσης, βλέποντας όλες τις ε, τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτές οι οποίες δεν μας φαίνονται τόσο ικανοποιητικές είναι εκεί όπου δεν θεωρείται αυτονόητο το ότι μιλάμε για εμπόριο. και όπου η προστασία οι συνθήκες διεξαγωγής του λιανεμπορίου μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι που μας ενοχλεί. Εμείς θέλουμε όμως, και το επεσήμανε και ο εισηγητής, ότι έχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, αθέμη του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να επιβάλλουν τις, ε, τους όρους τους, και των μικρότερων, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δεν έχουν την ίδια ευελιξία. Έτσι λοιπόν, Εάν κοιτάξουμε μόνο την υπόθεση αυτή από τη σκοπιά του ε, δικαίου του ανταγωνισμού, θα είναι πολύ μονομερής αυτή η θεώρηση. Αντίθετα, εγώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στο πώ θα κινηθούμε στην υπόθεση αυτή. Έχουμε δει λοιπόν μια σειρά από τροπολογίε, οι οποίε για μένα παρά είναι φιλελεύθερε, παρά είναι ε, ακραίε ω προ την ε, φιλελεύθερη θεώρηση και σημειώνουμε ότι δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε για άλλη μια φορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την σωστή λειτουργία του λιανεμπορίου. Um, Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούιλε. Κρίμα που δεν έχει έρθει ο κύριος Λούκερτ γιατί υπέβαλε κάποιες προτάσεις για διαγραφή που δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Εγώ θα ήθελα να υποβάλουμε έναν κανονισμό και για την δικαιόχρηση franchise και μιλήσαμε και γι' αυτό. Μπορώ να συμφωνήσω με την τροπολογία σας, αλλά ολοσχερή διαγραφή του άρθρου σε καμία περίπτωση δεν με βρίσκει σύμφωνη. Άρθρο 9. Σημαντικό και αυτό. Γιατί τα τοπικά καταστήματα είναι πολύ σημαντικά τα μικρά καταστήματα για την τοπική κοινωνία. Και είπαμε στην οδηγία για τις υπηρεσίες ότι θα πρέπει και οι τοπικές αρχές να μπορούν να λαμβάνουν μέτρα. Γιατί μιλήσατε για κάποιες ε, δομές και τις ε, μεγάλες υπεραγορές για, υπάρχει διαφορά μεταξύ του κέντρου των πόλεων και της περιφέρειας. Ε, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να πούμε ότι αντικαθιστά το ένα το άλλο. Έτσι λοιπόν ένας σχεδιασμός και από τις τοπικές αρχές θα ήταν χρήσιμος. Κατά τα άλλα, είπα και στην ε, τελευταία συζήτηση ότι είναι ισορροπημένη καλά αυτή η έκθεση. Έχει καλύψει σοβαρά θέματα ο κύριος Δε Ιόγκ και δεν έχουμε ιδιαίτερε παρατηρήσεις. Good. Uh, well, thank you very much. Perhaps um, I'll just pick up on my own reports. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που οι προτάσεις μου και οι ιδέες μου για την διεύρυνση των συνδέσμων με ε, μεταξύ της δικαιόχρησης franchise και των κανόνων ε, ανταγωνισμού είναι πολύ δόκιμη. Και θα το σχολιάσει και η συνάδελφος μετά θα μιλήσει για τις δικές της τροπολογίες, γιατί η δικαιόχρηση στο franchising είναι σημαντικό επιχειρησιακό μοντέλο, επιχειρηματικό μοντέλο και θα πρέπει όμως να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά γιατί μερικές φορές ε, περιορίζουν την ελευθερία των λιανεμπόρων ε, οι σχετικές διατάξεις. Όπως ε, μας επισήμανε και ο κύριος Βάπ, πολλές φορές γίνεται και πόλεμος τιμών μεταξύ των καταστημάτων. Η... Ε, το Amazon και το eBay και άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες πωλήσεων επίσης βρίσκονται σε διαφορετική θέση. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ θα υποβάλει και άλλες τροπολογίες. Ήδη έχει υποβάλει πολλές και συμφωνώ με ορισμένες από αυτές γιατί διευρύνουν αρκετά το πεδίο αλλά ο Κορνέλης ε, φαντάζομαι θα συμπηλήσει αυτές τις τροπολογίες και θα υποβάλει πολύ καλές συμβαστικές τροπολογίες που θα εμπλουτίσουν ε, και θα αναβαθμίσουν την έκθεσή του. Ας μην ξεχνούμε ότι έχουμε κάποιες ε, διατάξεις της πολιτικής ανταγωνισμού που ε, σχετίζονται με την πολιτική των κρατικών ενισχύσεων. Θα πρέπει να δούμε και εκεί την αλληλεπίδραση για να μην ε, ευνοηθούν ορισμένες επιχειρήσεις ή οργανώσεις αν και υπάρχουν σχετικές δυνατότητες από τα κράτη-μέλη που μερικές φορές είναι και εύλογες, αλλά μερικές χώρες προσπαθούν να, με παρεμβατικό τρόπο να ενισχύσουν τους ε, ντόπιου προμηθευτέ. Δεν είμαι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο είναι θετικό για την εσωτερική αγορά ή του καταναλωτέ, γιατί αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ευνοούμε του ε, καλούς ε, λιανεμπόρου και προμηθευτέ και να ενισχύουμε και το διαμεθοριακό εμπόριο, ανοίγοντα την αγορά και για νέου λιανεμπόρου. Και βλέπουμε τέτοια φαινόμενα όταν έχουμε κάποιον νέο προμηθευτή που εισέρχεται σε μια νέα αγορά, ιδιαίτερα στι καινούριε χώρε μέλη. Είναι όχι μόνο ο νέο αυτό ε, προμηθευτή ε, βοηθά και του ντόπιου και, και αναβαθμίζει τον ε, επαγγελματισμό του, αλλά ευνοεί το άνοιγμα και των δικών του αγορών προ του υπόλοιπου. Οπότε ουσιαστικά διευρύνονται οι δυνατότητε της αγοράς. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία λοιπόν και η ανάπτυξη του επαγγελματισμού της αλυσίδας ε, προμήθειας ό,τι αφορά την ποιότητα, την οργάνωση, την επεξεργασία, την συνεπή ε, αντίδραση, τη σωστή σήμαση και την ε, ετικετοθεσία. Όλα αυτά τα πράγματα με τη βελτίωση των συστημάτων πληροφορία και επικοινωνίας ουσιαστικά αναβαθμίζουν το ελληνικό εμπόριο και ευνοούν όχι μόνο τους καταναλωτές αλλά και το όλο σύστημα διανομής και την αλυσίδα διανομής. Και θέλουμε να βοηθήσουμε τους προμηθευτές να γίνουν πιο επαγγελματίες. Και από αυτή την άποψη χαίρομαι που καλύπτουμε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας, την αλυσίδα παροχή παροχής και δεν περιοριζόμαστε μόνο στα τρόφιμα, γιατί έχουμε και άλλες αλυσίδες ανεφοδιασμού και όχι μόνο των τροφίμων. Πάντως είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Κορνέλης Ντε Γιόγκ θα υποβάλει πολύ καλή πρόταση και θα λάβει μέρος και αύριο στη Στρογγυλή Τράπεζα για το Λιανικό Εμπόριο. Αυτά και περιμένω με ανυπομονησία και τις συμβαστικές αστροπολογίες. Ποιο άλλο θέλει το λόγο. Η κυρία Στάιλερ που έχει καταθέσει και τροπολογίε άλλωστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή και όλου όσοι έλαβαν το λόγο πολύ ευπρόσδεκτη εκθέση De Jong. Θα ήθελα απλώ να αναφερθώ σε μία-δύο από τις τροπολογίες μου. Την 66, ε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα τυπογραφικό σφάλμα στα αγγλικά, λέει third county και όχι third country, τρίτη χώρα δηλαδή και όχι κομιτεία. Αυτό είναι ένα τυπογραφικό ασφαλό σφάλμα. Θέλω να επιμείνω πάντως στο θέμα των τρίτων χωρών, διότι εκεί μπορεί να έχουμε το πιο ευάλωτο σε αθέμητες πρακτικές ε, κοινό και γι' αυτό θέλω ιδιαίτερα να επιμείνω στην πιο αυστηρή στάση εναντί στις τρίτες χώρες και βεβαίως θέλουμε μια αυστηρή αξιολόγηση της ε, εθελοντικής δέσμευσης η αναφορά σε έναν ε, διαμεσολαβητή που προτείνει ο κύριος Διόγκ, Ευρωπαίο διαμεσολαβητή για το θέμα αυτό, είναι χρήσιμη. Η πρωτοβουλία εν γέννη μου φαίνεται χρήσιμη και η στρογγυλή τράπεζα για το λιανεμπόριο που έχουμε για αύριο το απόγευμα θα είναι ασφαλώς ε, μια πλέον πηγή ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ. εάν θέλει η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κάποιος από την ομάδα της να μας κάνει κάποια σχόλια για τις τροπολογίες τότε. Επίσης την παρατήρησή σας ως προς την από, κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον μονομερή επιβολή μειώσεως ε, των τιμών θα πρέπει ο μηχανισμός ε, διαιτησίας ή ο μηχανισμός βέλτιστων ε, πρακτικών να φανούν χρήσιμοι, έτσι δεν είναι. Παρακαλώ την Επιτροπή. Ευχαριστώ, δεν έχω πολλά να συζητήσω. Θα δω και τις συμβαστικές τροπολογίες όταν έρθει η ώρα. Επί της ουσίας δεν έχω πάρα πολλά λοιπόν να παρατηρήσω, αλλά μια και έγινε ειδική αναφορά στο franchising. και έχοντας συζητήσει με τους συναδέλφους από το τμήμα ανταγωνισμού, το πρόβλημα για αυτούς, μπορώ να σας πω, δεν είναι η συνολική εξαίρεση, αλλά ξεπερνάει τους όρους της πολιτικής ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να ζητηθεί από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά τον κανονισμό για τους ε, ε, συνολικούς αποκλεισμούς. Για τις αθέμητες πρακτικές ε, ανταγωνισμού μπορώ να πω ότι αυτές ξεπερνούν ε, το θέμα του, της πολιτικής ανταγωνισμού και της συνολικής, ε, του συνολικού αποκλεισμού και θα ήθελα να επεκταθώ. Σε μια δύσκολη ερώτηση που διατυπώσατε για το ποια εθελοντική πρωτοβουλία θα μπορούσε κανείς να προβλέψει. Συνέπειες για τα όσα περιγράφεται και τα όσα ακούσαμε για τις κατοχώρες. Και χωρίς να θέλω να υποκαταστήσω τους αρμοδίους, που θα πρέπει να τοποθετηθούν, ξέρετε ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε τη Δευτέρα 16 του Πινούς Και αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει ή που αναμένεται για το επόμενο στάδιο είναι να ε, υιοθετήσουν την πρωτοβουλία αυτή οι εταιρείε. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε από σήμερα για μια τυπική προσφυγή ή διαμαρτυρία στους ε, διοικητές. Αλλά αν υπάρξει ζήτημα, ασφαλώς θα το αντιμετωπίσουμε. λόγο θα δούμε τις συνέπειες. Δεν πιστεύω όμως ότι είναι δυνατόν εγώ να δώσω εκτίμηση, πρόβλεψη για την έκφραση. Οι συζητήσεις αύριο με τη Στρογγυλή Τράπεζα θα είναι ασφαλώς πολύ χρήσιμες και αναμένω να τεθεί και πάλι το ζήτημα. Όταν θα έχουμε λοιπόν και την ομάδα των διοικητών, φαντάζομαι ότι κάποιος από αυτούς θα απαντήσει. Φαντάζομαι θα δώσετε και εσείς αύριο το παρόν. Θα συνεχιστεί λοιπόν η ζωή συζήτηση και αύριο για το ελληνικό εμπόριο. Και είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας ε, να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ελληνικό εμπόριο και τους λιανέμπορους γιατί είναι αναπόσπαστο τμήμα της εσωτερική αγοράς και μας ενδιαφέρει πολύ να το στηρίξουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Δηγιόγκ θέλει να προσθέσει κάτι. Έχουμε λίγο χρόνο πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω, Μάλκον. Όπως είπατε κι εσείς, η κυρία Κοράτσα Μπίλτ υπέβαλε πολλές τροπολογίες για την εσωτερική αγορά. Ε, πολύ συχνά είναι πολύ καλές οι προσθήκες αυτές. Άκουσα με πολύ προσοχή και τις παρατηρήσεις της κυρίας Γκέφχαρτ για την οδηγία για τις υπηρεσίες, την παροχή υπηρεσιών και έχει δίκιο, θα πρέπει να εγγύψουμε με μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα αυτά. Όπως είπατε, την επόμενη εβδομάδα θα συντάξω τις συμβαστικές τροπολογίες που θα εξετάσουμε με τους σχεώδεις ηγητές και προσβλέπω στη συνέχεια της συνεργασίας μας. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε προχωρήσει αρκετά γρήγορα. Ε, έχει έρθει η για το επόμενο θέμα, αλλά θα πρότεινα ε, να διακόψουμε για ένα δεκάλεπτο, γιατί κανονικά το επόμενο θέμα έχει προγραμματιστεί για τις 11 και 4. Και επειδή περιμένουμε και το επιτελείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους και οδησηγητές, ε, προτείνω μια σύντομη διακοπή, το πολύ δεκαλεπτά, ώστε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση του επόμενου θέματος στις 11 και 4 όπως είχε προγραμματιστεί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Uh, So, ladies and gentlemen, um, now that we have most of the shadow rapporteurs here. Ναι, και έχουν έρθει περισσότεροι και οδηγητές μας και η συγγήτριά μας η κυρία Βάιλερ ε, μέχρι τελευταία στιγμή γράφει τροπολογία θα την αφήσω να ολοκληρώσει τη σύνταξη και να καλωσορίσω τον Λουίς Φιλιπ Πιτσερά και τον Χαβιέρα Ριγκόη που ασχολούνται με το πακέτο αυτό και είναι συχνά καλεσμένοι στην Επιτροπή μας. κυρία Βάιλορ έχει ολοκληρώσει τις τροπολογίες της, έχει γράψει και την τελευταία. Σήμερα Έχουμε την τελική ανταλλαγή απόψεων για τι τροπολογίε και εξέταση των τροπολογιών πριν την αυριανή ψηφοφορία. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην συγγετριά μα μετά στην κυρία, στον κύριο Βαντεγκάμπ. Κυρία Ρούλερ και εγώ είμαστε εδώ, ο κύριος Μάντερς απουσιάζει, Όποιο άλλο θέλει το λόγο είναι ευπρόσδεκτο. Πρώτα όμω, ε, το λόγο έχει η συγγετριά μα, η κυρία Βάιλερ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για την ελαφρά καθυστέρηση η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι έλαβα μόλις μια νέα προφορική τροπολογία από τους φιλελευθέρους, τον οποίο έπρεπε να σημειώσω. Αλλά βέβαια ο αγώνας για ένα καλό αποτέλεσμα μας υποχρεώνει να συζητήσουμε τα πάντα. Δεν είναι λοιπόν τόσο σοβαρό το ότι κατατέθηκε τελευταία στιγμή τροπολογία. Ε, προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά, έστω και με κάποιες μικρές διαφορές σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ μικρές όμως, αλλά πιστεύω παρά τις μικρές αυτές ε, αλλαγές ότι έχουμε τον ίδιο αγώνα για τον καταναλωτή, για τη μικρομεσαία επιχείρηση και για την προστασία του βιομηχανικού κλάδου και έτσι νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια καλή και καλά ισορροπημένη πρόταση για αύριο. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα θέματα που είχα εκθέσει στην προηγούμενη συζήτηση. Παραμένουμε στην αυτή γραμμή. Έχουμε αλλάξει τον ορισμό το πεδίο εφαρμογή. Και πιστεύουμε ότι το ράδιο φάσμα είναι πόρος ο οποίος μπορεί να αξιοποιείται όλο και περισσότερο και με τρόπο όλο και πιο αντισυμβατικούς. Σε αυτό θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Θέλουμε να συμφωνήσουμε στο Συμβούλιο ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση. Και για να περάσω στα ιδιαίτερα μας μελήματα για την ε, νέα μεταρρύθμιση, για τους φορτιστές, chargers, στην προφορική τροπολογία που είδαμε τώρα και λόγω των όσων μας επεσήμαναν οι διάφοροι συνάδελφοι στο θέμα αυτό, η ιδέα ενός κοινού ε, φορτιστή, universal charger, οικουμενικού, δεν μπορεί βέβαια να είναι ένας φορτιστής ο οποίος θα ισχύει για, όλα τα, ε, για όλες τις συσκευέ, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ιδιαίτερες κατηγορίες ε, για τα προϊόντα, για κάποια προϊόντα, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό είναι στα κινητά τηλέφωνα να έχουμε έναν φορτιστή και θα πρέπει να δεσμευτεί ο κλάδος να ε, προσφέρει στον καταναλωτή φορτιστές συμβατούς με τις διάφορες συσκευές. Στην κινητή τηλεφωνία κυρίως. Πάντως, στην φράση «ο φορτιστής μπορεί να πωλείται χωριστά», εγώ θα ήθελα να τη διαγράψω τη φράση αυτή, γιατί μου φαίνεται τόσο αυτονόητη. Το είπα στους συνελευθέρους μόλις τώρα, ότι αν ε, βγει αυτό το πράγμα πιο έξω, θα μας ε, γελιοποιήσουν ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωση άμα φανεί ότι λέμε «Α, πρέπει να πωλείται χωριστά ο φορτιστής». Μα είναι αυτονόητο. Αν κάποιος έχει ένα φορτιστή με τη συσκευή αγοράσει ε, ή λάβει μάλλον και τον χάσει, θα πρέπει να μπορεί να πάει να αγοράσει ένα καινούριο. αυτονόητο λοιπόν. Μάλκολμ, μία-δύο ε, τροπολογίες σου θα χρειαστεί να απορρίψω διότι θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητες και μπορεί να οδηγήσουν σε αβεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα. 105, Μάλκολμ. Πληροφορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με το, με το του ραδιοφάσματος και τις οποίες θεωρώ απαραίτητες για τις αρχές μας. Ε, την 105 λοιπόν δεν τη δέχομαι, δέχομαι όμως την 103 εκεί που γίνεται Ε, η αναφορά στο όπου είναι δυνατόν, γιατί αυτό το είχατε πει προφορικά αν δεν απατώμε, γιατί η Επιτροπή λοιπόν δεν δέχεται να ε, δεν δέχεται την ε, τροπολογία αυτή, το να υπάρχει ενσωματωμένη ορθόνη και να μπορεί να πληρούνται αυτή η υποχρέωση μέσω λειτουργία που επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει την εμφάνιση των απαιτούμενων πληροφοριών. Το ότι είναι δυνητική η διατύπωση και δεδομένου ότι θεωρώ ότι μάλλον την Αγγλία εννοείται ιδιαίτερα, ότι εκεί θα πρέπει να καθίσταται δυνατή αυτή η προσφορά. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο να δεχθούμε. Στην 116 και τη δυνατότητα για προσφυγή του καταναλωτή για προϊόντα που δεν ε, συμμορφούνται είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω. Νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να το εισαγάγουμε. Γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη θέση στην οποία να μπορεί να απευθυνθεί ο καταναλωτή. ο πολίτης. Ε, στη Γερμανία, παραδείγματι, δεν υπάρχει αρμόδια αρχή, δεν θεωρούν ούτε οι αρχές, η αρχή τηλεπικοινωνιών, ούτε καμιά άλλη αρχή ε, ότι είναι αρμόδιες για να δέχονται τέτοιου είδου ε, διαμαρτυρίε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ρυθμιστεί πλέον. Αυτά. Νομίζω ότι έτσι εντάσσουμε το κείμενο αυτό και στη γενικότερη δέσμη της κυρίας Ρόιτοβα και ολοκληρώνουμε το πακέτο ε, και με αυτό το κομμάτι της δικής μου εκθέσεως. Στα υπόλοιπα δεν έχουμε ιδιαίτερες ε, αλλαγές εσείς με τα προηγούμενα, με τόσο είπαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Αύριο ίσως ε, με την ψηφοφορία θα επισημάνω, αλλά σας το λέω και τώρα, ότι θα ήθελα όπου είναι δυνατόν ή όπου μπορούμε να επιβίνουμε. Κύριε Σφαμ, με ακούτε όπου μπορούμε να επιμείνουμε ή να αποπειραθούμε έστω να επιμείνουμε και να πιέσουμε, να επιδιώξουμε τα κράτη-μέλη, να πιέσουν και αυτά από πλευρά του. το ταχύτερο δυνατό να εγκριθεί, να προχωρήσει δηλαδή η διαβούλευση για να εγκριθεί το πακέτο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε κάποια ενημέρωση ότι κατά πάσα πιθανότητα τα κράτη-μέλη δεν υπολογίζουν να κλείσει το πακέτο αυτό μέσα στην τρέχουσα θητεία, πράγμα το οποίο εμένα θα με λυπούσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βαντεκάπα έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, με την κυρία Βάιλερ ξέρω, πάντα οι φιλελεύθεροι φταίνε. Να συνεχίσω στα Ολλανδικά, να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια ε, για την ενέργεια με την οποία χειρίζεται αυτό το φάκελο και για την ε, επιμονή της. Ε, Γενικώ συμφωνούμε με τις ε, τροπολογίες και την προσέγγιση. Είναι ένας από τους φακέλους, Πρόεδρε, που δεν αφορά την ελευθερία του τύπου, ούτε ευρύτερα την πολιτική αυτή, αλλά είναι πολύ σημαντική για την εναρμόνιση αυτού του εξοπλισμού στην Ευρώπη και ε, επιφέρει και εξοικονόμηση πόρων. Οι τροπολογίες και η προφορική τροπολογία για τους φορτιστές. Σε αυτό το ζήτημα συμφωνώ. Στα όσα λέει η νομίζω ότι υπάρχει σωστή προετοιμασία του φακέλου ε, και ε, σύνδεση του με τους φακέλους του κυρίου Ρόιτοβα και ελπίζω του αύριο να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Δυστυχώ εγώ προσωπικά δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ, όμως έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυρία Βάιλερ και σε εσά στην ιδιότητά σας ως σκιώδου. Ευχαριστώ πολύ. Okay. I'm, I'm afraid I... Δυστυχώς ούτε εγώ θα είμαι αύριο εδώ, αλλά θα είναι εδώ αντιπρόεδρος. Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει η πρόταση τη κυρία Βάιλερ. Όμω, οι συνάδελφοί μου θα με εκπροσωπήσουν. Ο κύριος Μάντες δυστυχώς ε, λείπει, αποσιάζει. Η κυρία Ρούλε νομίζω έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Υποστηρίζουμε την ε, πρόταση της προτάσης της κυρίας Βάιλερ και θα το εκφράσουμε και την ψηφοφορία αύριο. Ναι. Ξέρω ότι είστε από τους είναι συνεπείς, είστε πιο συχνά εδώ. Να σχολιάσω κάποια από τα δικά μου σχόλια, τις τροπολογίες στην ιδιότητά μου ως ε, σκιώδους. Να ευχαριστήσω αρχικά την κυρία Βάιλερ ε, που πολύ επικοινωνικά αποδέχθηκε σημαντικό ρυθμό τροπολογιών μου. Δεν ήμουν απολύτως σαφής ε, όμως. Από ό,τι κατάλαβα, δεχθήκατε την πρότασή μου για την ηλεκτρονική σήμανση, γιατί έχουμε υποβάλει περαιτέρω πληροφορίες γι' αυτό. Αν θυμάστε, το συζητήσαμε για την προηγούμενη φορά. Και η Επιτροπή διευκρίνησε ότι υπάρχει αδυναμία των αρχών επιτήρησης της αγοράς να ελέγξει ε, εξοπλισμό όταν δεν ε, αναγράφεται η λειτουργία της μπαταρίας στην οθόνη. Όσοι έχουν αγοράσει ένα καινούριο ε, κινητό Ξέρετε ότι σε τέτοιου είδους τηλέφωνα πάντα υπάρχει ένα πλαστικό ε, κάλυμα της οθόνης και ε, λέει η αγορά λοιπόν ότι αυτό το τμήμα της συσκευασία θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Κάτι άλλο. Μπορείτε να ελέγξετε αν είναι μοντέρνο και σύγχρονο αυτό το κινητό που έχετε αν δείτε στο πληκτρολόγιο και πληκτρολογήσετε, μισό λεπτό να ανοίξω και εγώ το δικό μου. Στο πληκτρολόγιο λοιπόν, αν βάλετε ε, αστερακι δύο, 07 δίωση και ε, καλέσετε, θα δείτε αυτή την οθόνη ο, του θαύματος. Και στην Apple θα το δείτε αυτό. Τέλος πάντων, είναι ένας ε, συνήθις ε, κωδικός που αν τον πατήσετε θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η κυρία Στάιλερ, παίζετε πριν με το κινητό σας, μπορείτε να δείτε αν και το δικό σας είναι εξίσου σύγχρονο με το δικό μου. Βλέπω ότι όλοι τώρα θέλετε να δείτε το κινητό σας, να δείτε αν λειτουργεί. Λοιπόν, αστεράκι, δίεση, 07 δίεση. και θα σας πάει απευθείας σε, αυτή, αυτή την οθόνη με αυτές τις πληροφορίες. Αν έχετε iPhone 5. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, ε, αυτή η νέα πρόταση είναι αρκετά εποφελής. Είναι και κάτι που θα πρέπει να επιδιώξει και το Κοινοβούλιο. Γιατί προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, προς τέτοια κινητά και η πρόσβαση των καταναλωτών στις πληροφορίες είναι πολύ σημαντική γιατί αλλιώς ε, θα μπορούσα να το είχα πετάξει και αυτό μαζί με την υπόλοιπη συσκευασία σε ό,τι αφορά του γενικού όρου χρήση και το καθεξή. Χαίρομαι λοιπόν που το αποδεχόμαστε. Μια άλλη γενική παρατήρηση. Βάσει και τη προσέγγιση της κυρίας ε, Βάιλερ, την τροπολογία 118 σε αντίθεση με την 120 πρέπει να το ψηφίσουμε. Αλλά προφανώ ε, είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να υπάρξουν πραγματεύσει με το Συμβούλιο σε μεταγενέστερο στάδιο. Και έχω δει και προφορική τροπολογία του κ. Μάντας για αυτούς του οικομανικούς ε, φορτιστές, Universal Chargers, που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί πρέπει ε, πράγματι και εμείς ε, να στηρίξουμε με κάποιον τρόπο αυτό το είδος φορτιστών στην πρότασή μα. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να στηρίξουμε κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώ στηρίζουμε ω Επιτροπή. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε σε συμβιβασμό σπιτού του και μετά έχω κάνει και αρκετές λεπτομερείς προτάσεις. Τα περισσότερα τα δεχθήκατε σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες και τη σήμανση. Είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης ε, ευθυγράμμιση και με την ακριβή διατύπωση και συμμόρφωση με το νέο ε, κανονιστικό πλαίσιο, όμως αυτό σίγουρα θα συμβεί στη συνέχεια. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο για το ραδιοξοπλισμό. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε αν έχουν άλλες παρατηρήσεις εν ώψη της αυριανής ψηφοφορίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε ό,τι φορά κάποια ζητήματα διατύπωσης μπορούμε να τα εξετάσουμε στη συνέχεια, όμως ας ε, εστιαστούμε σε τέσσερα σημαντικά για μας ε, θέματα, όπου ακόμα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Πρώτον, για το πεδίο στο φάσμα. Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, πρόθεσή μας ήταν να επικεντρωθούμε στους ε, αναμεταδότες, transmitters και μόνο. Ε, μπορούμε να δεχθούμε και ως ε, εναλλακτική να αποδεχθούμε και τους δέκτες, receivers. Υπάρχει όμως ακόμα ένα πρόβλημα στο πλαίσιο της ε, επικοινωνία, της κοινοποίηση ε, τέτοιου εξοπλισμού. Γιατί θεωρούμε ότι ε, όλος ο εξοπλισμός που εκπέμπει κύματα και μπορεί να έχει παρεμβολές με το φάσμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογή της νομοθεσίας. Αν λοιπόν εισαγάγουμε τον όρο communication δεν θα ισχύει αυτό. Δεύτερον, για το Μητρό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό εργαλείο ε, για τις ε, αρχές επίβλεψης της αγοράς. Ε, για χρόνια εξετάζουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία αυτών των αρχών. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για εξαιρετικές συνθήκες και περιστάσεις. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει άχθος για τον κατασκευαστή σε ό,τι φορά αυτό το μητρό. Επομένως, ε, θεωρούμε ότι σε πολλές χώρες, ε, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, εκεί λοιπόν αυτό το μητρό είναι υποχρεωτικό. Ανεξαρτήτως ε, του τι λένε οι αρχές αυτές. Λοιπόν, για την ηλεκτρονική σήμανση και εμεί θεωρούμε ότι δεν πληρούνται ακόμα οι προϋποθέσεις για να ακολουθήσουμε και να κινηθούμε προς την ηλεκτρονική αγορά, την ηλεκτρονική σήμανση μάλλον. Ε, τώρα, για να έχουμε αυτό το αυτοκόλλητο στην ε, ε, οθόνη, κάποια από, αυτά τα σήματα θα έχουν τέτοιο σήμα στον εξοπλισμό, όπως το C-marking. Επομένως, πέραν της φόρτισης του εξοπλισμού υπάρχει και το ζήτημα ε, των αρχών επιτήρησης της αγοράς που κάποιες φορές ελέγχουν 10-20 προϊόντα. Επομένω, εάν κάθε φορά πρέπει να βγάλουν το προϊόν από τη συσκευασία, να το συνδέσουν, να, το θέσουν σε λειτουργία για να δουν εάν υπάρχουν οι προβλεπόμενες ενδείξεις, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι δύσκολο να εφαρμοστεί πρακτικά. Βεβαίω, η ηλεκτρονική σήμανση είναι μια κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε, το έχουμε ξαναπεί, όμως ε, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά για να γίνει αποδεκτό στην νομοθεσία. Λοιπόν, για τους οικονομικούς ε, φορτιστές, εκπονούμε μελέτη για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της εφιστάμενης εθελοντικής συμφωνίας για τα κινητά τηλέφωνα. Η μελέτη αυτή καλύπτει και άλλες μικρές ηλεκτρονικές συσκευές σε αυτόν τον κλάδο. Με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θέλουμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη δυνατή κατεύθυνση. Βεβαίω αναμφίβολα κινούμαστε προς τους οικομενικού φορτιστέ. Το θέμα είναι πώς, ε, ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση σήμερα. Να συνεχίσουμε με την εθελοντική Συμφωνία ή να προβλέψουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Από δική μα πλευράς δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να ε, ξεκαθαρίσουμε ποια επιλογή προτιμούμε. Εάν το συμπεριλάβουμε στην οδηγία, σίγουρα θα προτιμήσουμε τρομοθετική προσέγγιση. Θα προτιμούσαμε λοιπόν να γίνεται αναφορά ε, ως προς αυτό σε μια ιταλογική σκέψη και έτσι το έχουμε, έχουμε συμπεριλάβει στην πρότασή μας τη δυνατότητα νομοθέτησης περί των φορτιστών μικρών ηλεκτρονικών συσκευών στο μέλλον βάσει των συμπερασμάτων ε, σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση και τις υφιστάμενες ανάγκες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, Mrs. Weiler, did you want to, um... Σας ευχαριστώ. Κυρία Βάιλερ, έχετε άλλα σχόλια. Ναι. Δεν θα κάνω νέα σχόλια, διότι γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιφυλάξεις της Επιτροπής ήδη. Την έχω δει και σε ε, προσωπικές ε, συνομιλίες Νομίζω ότι απλώς καταλήγουμε σε διαφορετικές διαπιστώσεις. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο, πώς θα τοποθετηθούν και πώς, τι είδους αντιπαράθεση θα αναπτυχθεί μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Και έως εκ τούτου εγώ θα πρότεινα να παραμείνουμε στη γραμμή που έχουμε ορίσει για τις ε, ψηφοφορίες μας και μόνο για τις τροπολογίες 103 και 111. Παρακαλώ αγαπητέ Μάλκομ, συζητήσετε με την Επιτροπή. Η Επιτροπή μας ε, επιμένει ότι τάσατε κατά των τροπολογιών γιατί θεωρία ότι στην πράξη δεν θα είναι εφαρμόσιμες. Εγώ νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε κάποια λύση στη διαπραγματεύση μαζί τους. Για τα υπόλοιπα ευχαριστώ πολύ για την ε, θετική στάση. Ο Επίτροπος Σταγιάννη μάλιστα έχει εκφράσει τη μεγάλη του χαρά και ικανοποίηση για την επιτέλους ε, κατάθεση της, πρώτης της νομοθετικής πρότασης. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι περίμενα πιο θετική ακόμα στάση. Και βλέπουμε όλοι δυστυχώς ότι πολλές φορές η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών μας λέει ναι, ναι, ναι, θα το κάνουμε, θα το αναλάβουμε, θα δεσμευθούμε», αλλά δύο χρόνια μετά τελικά καταγγέλει τις δεσμεύσεις αυτές και δεν τις υλοποιεί. και χαίρομαι που επιτέλου έχει ε, η Επιτροπή και πάνω από ο Επίτροπος ταχθεί υπέρ αυτής της ε, υποχρέωσης, υπέρ αυτής της τοποθέτησης στο νομοθέτημα. στο, στη διαπραγμάτευση μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε υποχωρήσει σε κάποια λιγότερο κρίσιμα σημεία, αλλά το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επιμείνουμε. Ωραία, ευχαριστώ για την ε, υποστήριξή σας από ό,τι ξέρω εγώ, ήδη υπάρχουν κάποια ε, μέτρα όπως ε, στην, σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, ε, η Ιαπωνία. Ακόμη και οι ΗΠΑ το σκέφτονται για το ηλεκτρονικό σήμα. Ελπίζω να μην μείνουμε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε είναι λογικό για τις ε, νέες συσκευέ και τον νέο εξοπλισμό που θέλουμε να κυκλοφορεί. Ίσως ε, ε, μπορούμε να βρούμε μια διατύπωση. Και ε, θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό σε σχέση με το προστατευτικό αυτό πλαστικό φύλλο που υπάρχει πάνω στις συσκευέ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο. Και πάλι ήμασταν πολύ διεκπαιρωτικοί και αποτελεσματικοί. Και πάλι έχουμε τελειώσει λίγο νωρίτερα. Βέβαια έχει έρθει η συγκήτρια για το επόμενο θέμα, αλλά να δούμε αν έχουμε απαρτία των σκιωδών εισηγητών και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπω τον κύριο Παντσέρη, αλλά δεν βλέπω τον κύριο Κρόιτσμαν και τον κύριο Μπιέλαν. Αλλά βλέπω τον κύριο Κάρνεγκη από τη Γενική Διεύθυνση εσωτερική Αγοράς. Perhaps we'll just Ας κάνουμε μια ολιγόλεπτη διακοπή για να μαζευτούμε όλοι. Και η βοηθή παρακαλώ να καλέσω τους πιο δυσηγητές για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω αν θα έρθει και ο κύριος Άγκστρομ για τους πράσινους. Πέντε λεπτά διακοπή. Για να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα από το προβλεπόμενο.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 Uh, λοιπόν, συνάδελφοι, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε απαρτία των σκιωδών εισηγητών και της εισηγήτρια φυσικά. Καλωσορίζω την κυρία Μπάστο, που είναι η εισηγήτριά μα για την γνωμοδότηση που θα επιδώσουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και μάλιστα είναι μεικτή γνωμοδότηση για δύο σημαντικές αναθεωρήσεις. Η μία αφορά ε, την ε, κοινοτική νομοθεσία για το ευρωπαϊκό σήμα και η δεύτερη είναι μια αναδιατύπωση για την νομοθεσία των κρατών μελών περί Είναι σημαντικό να δώσουμε τις γνωμοδοτήσεις αυτές ε, το πρίσμα της δικής μας Επιτροπής και θα μπορούσε στο μεταξύ να μας ενημερώσει η κυρία Μπάστος για τις σχέσεις της και τις συνεννοήσεις που κάνει με την αρμόδια καθήλια επιτροπή, την νομική επιτροπή. Είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα ακούσουμε την παρουσίαση από την εισηγήτρια. Μετά έχουμε τον κύριο Παντσέρη και όδη από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, τον κύριο Χατζημαρκά και που αντικαθιστά τον κύριο Κρόσμα, Ο κύριος Άγκστρομ δεν έχει έρθει ακόμη, ο κύριος Μπιέλαν ε, επίσης ε, είναι στο δρόμο. Και καλωσορίζω και τον κύριο Κένιγκ που θα παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, λοιπόν, δίνω το λόγο στην κυρία Ρεζίνα Μπάστος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλημέρα σας. Είναι για μένα ιδιαίτερο προνόμιο ε, η σύνταξη της γνωμοδότησης, το δύο γνωμοδοτήσεων για το κοινοτικό σήμα και την ομοθεσία των κρατών μελών περισημάτων αναδια εκτύπωση. Τα εμπορικά σήματα έχουν τεράστια οικονομική αξία στην εσωτερική αγορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η νομοθετική αυτή αναθεώρηση είναι απαραίτητη, μια και θέλουμε να τονώσουμε την εσωτερική αγορά, να την ενισχύσουμε, να προστατεύσουμε τα εμπορικά σήματα και πάνω απ' όλα να καταπολεμήσουμε την απομίμηση, την πειρατή και τι ε, παραποίησει. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ε, έχει διάφορου στόχου. Καταρχήν προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης ε, καθιστώντας πιο προσιτό το σύστημα των εμπορικών σημάτων και πιο αποτελεσματικό για τις επιχειρήσεις με μείωση του κόστους και μείωση των διατυπώσεων και αύξηση της ασφάλειας δικαίου. Άλλος στόχος είναι να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών Ινστιτούτων ε, και Οργανισμών των Κρατών Μελών και του ε, Ινστιτούτου Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς προκειμένου να προωθηθούν ε, οι βέλτιστες πρακτικές. Τρίτος στόχος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η προσαρμογή του κανονισμού στη συνθήκη της Λισαβόνας και την ανάγκη αντιμετώπιση του θέματος των κεντρικών οργανισμών. Σίγουρα το εμπορικό σήμα δημιουργεί πολλά ωφέλη για τις επιχειρήσεις και συμβάλλει ταυτόχρονα στην προστασία των καταναλωτών. Η προστασία των εμπορικών σημάτων ε, είναι αυτονόητο ότι μειώνει το κόστος ε, για τους καταναλωτές, εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ε, για το προϊόν και επίσης βελτιώνει τις επενδύσεις προς καινοτομίες. Βέβαια, ο κύριος εχθρός του εμπορικού σήματος είναι η πειρατεία, η απομίμηση και οι παραποίησει, γιατί δημιουργούν προσκόμματα στις, στην καινοτομία, παραβλάπτουν την ανταγωνιστικότητα, καταστρέφουν θέσεις απασχόλησης, ε, πλήττουν τα δημόσια οικονομικά, εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη και σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα απειλούν ε, την προστασία και την ασφάλεια των ε, Ευρωπαίων καταναλωτών. Η ιστορία του εμπορικού σήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακροχρόνια αλλά συνεπής. Έχουμε ήδη 15 χρόνια που εφαρμόζουμε το κοινοτικό σήμα με πολύ σταθερές βάσεις και μάλιστα κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερα αιτήματα και το Ινστιτούτο για την Εναρμόνιση της Εσωτερικής Αγοράς για να σας δώσω ένα εύγλωτο παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας του εμπορικού ε, σήματος είναι το 2011 έλαβε την χιλιοστή αίτηση από την έναξη της δραστηριότητά του το 1997. Το σύστημα των εμπορικών σημάτων στηρίζεται στην αρχή της συνύπαρξης και της συμπληρωματικότητα μεταξύ της προστασίας των εμπορικών σημάτων σε ε, εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ θετική λοιπόν η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμφωνούμε ότι δεν έχουμε ανάγκη για σημαντικές ε, και ρηξικέλευθες ε, μεταρρυθμίσεις, γιατί οι βάσεις που διέπουν και τα θεμέλια που διέπουν το εμπορικό σήμα είναι έγκυρες, Οπότε χρειαζόμαστε έναν εξυγχρονισμό σωστά στοχοθετημένο, ώστε να έχουμε πιο εύκολη, αποτελεσματική και φθηνή προστασία των εμπορικών σημάτων. Έτσι θα ενισχύσουμε την καινοτομία, θα προσεγγίσουμε επενδύσεις, θα δημιουργήσουμε νέα αγαθά και υπηρεσίε και θα ανταποκριθούμε στι ε, νέε ανάγκε των καταναλωτών και φυσικά στην ανάγκη επενδύσεων και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής θέλει να βελτιώσει το νομοθετικό πλαίσιο και να αυξήσει ε, τους βαθμούς, το βαθμό προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, διευκρινίζει το καθεστώς που ισχύει για τα προϊόντα διαμετακόμιση, ένα πολύ ευαίσθητο σημείο της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα και επίμαχο, δεν υπάρχει συμφωνία γι' αυτό, προσθέτει σημαντικές καινοτομίες όπως είναι ο ορισμός του του σήματος και κάποιες ευκρινήσεις ε, για την προστασία ε, παραδοσιακών προϊόντων ή ενδείξεων ε, γεωγραφίας προέλευσης. Η δική μου γνώμη τώρα, ως εισηγήτρια των ομοδοτήσεων, είναι υπέρ της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποβάλλω κάποιες προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πρώτη τροπολογία αφορά την ενίσχυση του ρόλου των εθνικών αρχών στο σύστημα προστασίας των σημάτων και στην καταπολέμηση της παραποίησης και απομίμησης. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, το διεθνές εμπόριο ε, με παραπημένα προϊόντα έχει αυξηθεί κατά 100 ε, δισεκατομμύρια το 2000 από σε 50 δισεκατομμύρια το 2007 και μάλιστα οι αξίες, οι, οι τιμές που προτείνονται και τα στοιχεία για τις εθνικές τελωνιακές αρχές διαπιστώνουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερα παραπημένα προϊόντα. έχει αυξηθεί τα κατασκευθέντα παραπημένα προϊόντα κατά 70% τα τελευταία πενταετία, κάτι που κρούει το κόδωνα του κινδύνου. Επίσης θέλουμε να διατηρήσουμε την δυνατότητα ε, κατάθεσης ε, του αιτήματο για κοινοτικό σήμα είτε στις ε, στα Εθνικά Ινστιτούτα Προστασίας του Σήματος είτε στο, ε, στο κοινοτικό, προκειμένου να γίνει πιο προσιτό το σύστημα και να μην δίνεται αίσθηση στους Ευρωπαίους πολίτες ε, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ε, είναι πολύ μακριά από αυτούς. Θέλουμε να κρατήσουμε την αρχή της εγκύτητας σε ό,τι αφορά τι ε, υπηρεσίε, οι οποίε μπορούν να αποτείνονται οι Ευρωπαίοι πολίτε. Γιατί οι πολίτε όλο και περισσότερο θεωρούν ότι οι Βρυξέλλε βρίσκονται πολύ μακριά από αυτούς. Η τρίτη τροπολογία που προτείνω αφορά την ε, ανάλυση των, ε, της επιχειρηματολογίας για την απόρριψη της αίτησης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε την ε, νομολογία έχει, να μην έχουμε μόνο τους απόλυτους ε, λόγους. Θέλουμε να διατηρήσουμε το σύστημα όπως έχει, γιατί ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελαφρύνει το κόστος επιτήρησης. Ε, επίσης, εμποδίζει τη δημιουργία συγκεκριμένων σημάτων, περιορίζει τις παραβιάσεις, αλλά και ελαφρύνει το φόρτο των δικαστηρίων, περιορίζοντας τις ε, διαφορές. Μάλιστα αυτό το σύστημα ήδη ισχύει σε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τέταρτη τροπολογία μου αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού που θα πρέπει να απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος ε, της σύνθεσης αυτής είναι να εξασφαλιστεί μια θεσμική ισορροπία και να επιτραπεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η αποτελεσματική συμμετοχή του στην εποπτεία του οργανισμού. Επέμπτη τροπολογία αφορά τα νέα καθήκοντα του οργανισμού. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να αναθέσουμε νέε αρμοδιότητε στον οργανισμό, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη διαχείριση και την προώθηση των ονομασιών προέλευση των ή των προστατευμένων γεωγραφικών ενδείξεων θα μπορεί επίσης να προωθεί και να διαχειρίζεται άλλα σημαντικά δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία με βάση το άρθρο 118 της συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία άλλη τροπολογία, η έκτη, θεωρεί σκόπιμο ο οργανισμός ε, να ασκεί και κάποιες υπηρεσίες ε, διαμεσολάβησης ε, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων σε προαιρετική βάση μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων. Έβδομη τροπολογία, μείωση των τελών. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει τα επίπεδα των τελών για να μειωθεί το κόστος γιατί όταν υπάρχει ένα πλεόνασμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ε, για μέτρα και σχέδια για τη βελτίωση του συστήματος εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει όταν δημιουργείται τέτοιο πλεόνασμα ε, που θα επιστρέφει στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Προτιμώ να μένουν αυτά τα πλεονάσματα στον οργανισμό και να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση του συστήματος. Να μην υπάρχει μεταφορά προς τον κοινοτικό προπολογισμό. Επίσης τα πλεονάσματα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις νέες αρμοδιότητες που πιστεύω θα πρέπει να ανατεθούν στον οργανισμό για να βελτιωθεί το σύστημα. Ε, το κείμενο, ακριβώς επειδή έχει πολλούς περιορισμούς τη αφορά την ε, έκθεσή του, αποφάσισα να υποβάλω ξεχωριστές τροπολογίες για να το διαβρύνω και να το εμπλωτίσω. Θέλω πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, να ενισχύσω τον έλεγχο της προστασίας ε, των εμπορικών σημάτων, αλλά ε, και να προωθήσουμε και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα ζήτημα που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους καταναλωτές. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Γι' αυτό και θα πρέπει να είναι και αξιόπιστο. Θα, θα, θα πρέπει οι καταναλωτές να μπορούν να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο όντας βέβαια για την αξιοπιστία του. επίση ε, το σήμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται και από το ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί το ηλεκτρονικό εμπόριο εξασφαλίζει την ανωνυμία και κάνει πιο, ελαστικό, πιο ελαστική την αγορά. Οι επιχειρήσεις όμως και οι καταναλωτές ε, δεν ε, θα πιστούν αν θέλουμε να κάνουμε πιο αυστηρές ε, τις διατάξεις για το κλασικό συμβατικό εμπόριο και εξαιρέσουμε από τους αυστηρότερους αυτούς ελέγχους ε, το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα μένει ανεξέλεγκτο. Κάτι τέτοιο δεν θα βρει σύμφωνα ούτε τις επιχειρήσεις ούτε τους καταναλωτές. Διάβασα πολλές ε, τροπολογίες για τις παραποιήσεις και απομιμήσεις κάποιων προϊόντων που προστατεύονται από εμπορικό σήμα δεν θέλω να, αναφέρουμε συγκεκριμένα σήματα ή συγκεκριμένες ε, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συγκεκριμενε πλατφορμες ηλεκτρονικου ή περιπτωσει οπου η προστατευμένων προϊόντων που τίθενται σε εμπορίες σε συγκεκριμένε πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου ε, σε ορισμένες χώρε ε, φτάνουν σε τάξη μεγέθους 40%. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τον έλεγχο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Άλλη τροπολογία μου αφορά τη σύνθεση, επαναλαμβάνω, του Διοικητικού Συμβουλίου ε, του Οργανισμού. Προσθέτω εκεί έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σε ό,τι αφορά την ε, επιλογή του εκτελεστικού διευθυντή, προτείνω κάποιε αλλαγέ. Δεν θα πρέπει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει του υποψηφίου, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή προεπιλογής που θα παρτίζεται από δύο εκπροσώπους ε, των κρατομελών, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά την απόφαση για την ανάκληση του εκτελεστικού διευθυντή θα πρέπει να λαμβάνεται η απόφαση με πλειοψηφία δύο τρίτων και όχι απλή πλειοψηφία. Επίσης, η πρόταση θα μπορεί να εκπορεύεται είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην έχει αποκλειστική πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση αυτή. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία ενός κέντρου διαμεσολάβησης και διατησία, προκειμένου το σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό, λιγότερο επαχθές και απλούστερο και πιο ευέλικτο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι περιμένω στις ε, προτάσεις των σχεδόν εισηγητών και πιστεύω ότι από κοινού θα καταλήξουμε σε έγκαιρο και καλό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να τηρήσουμε, το οποίο πιστε, προβλέπει προθεσμία ε, για τις τροπολογίες 20 16 ε, Σεπτεμβρίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι, 14 Οκτωβρίου εξέταση και 5 Νοεμβρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή. Και ελπίζω με τις γνωμοδοτήσεις μας να συμπληρώσουμε την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ και περιμένω τους σκιώδεις συγγητές και τις παρατηρήσεις τους. Καλώς ευχαριστώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο βεβαίως. Φαντάζομαι ότι θα δώσουμε θα κάνω την προσπάθεια που χρειάζεται οι συγγητέ. 5 Νοεμβρίου νομίζω τώρα έχει πάει η ημερομηνία. Ας ακούσουμε λοιπόν τους σκιώδη με τον κύριο Παντσέρη πρώτο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σύντομα θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω τη σημασία της, ε, της δέσμης μεταρρυθμίσεων που μας έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοβουλίες οι οποίες ασφαλώς θα περιορίσουν το κόστος, θα καταστήσουν πιο αξιόπιστο και προβλέψιμο το σύστημα καταχώρηση σημάτων. Είναι, πιστεύω, μία μεταρρύθμιση χρήσιμη, μια μεταρρύθμιση που βελτιώνει τις συνθήκες στην αγορά και, την, ε, και προστατεύει περισσότερο από την απομίμηση και κυρίως προϊόντα απομίμησης που περνούν σε διαμετακόμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικά μας προϊόντα και σήματα. Η πρόταση λοιπόν της κυρίας Μπάστος είναι ακριβώς, επιδιώκει ακριβώς αυτό το στόχο, υποστηρίζω τις τροπολογίες της, οι οποίες ιδιαίτερα στόχο έχουν να προστατεύσουν το κοινοτικό σήμα σε προϊόντα που ε, είναι σε καθεστώς διαμετακόμισης. Ζητούμε λοιπόν από την αρμόδια υπηρεσία να διαχειρίζεται τα σήματα και τις ονομασίες προελεύσεως και τα λοιπά σήματα που μπορεί να περιλαμβάνονται ε, να καλύπτονται μάλλον από το σήμα. Ωστόσο θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε στο νομοθέτημα αυτό την προστασία των καταναλωτών, που είναι ιδιαίτερο μέλημα της Επιτροπής μας και θέλω να επιμένω στα εξή. Πρώτον, θέλω να υπενθυμίσουμε και να ενισχύσουμε τον παραδοσιακό ρόλο της, του σήματος, της επιχείρησης του κοινοτικού σήματος. Ο ουσιώδης ρόλος του σήματος είναι να δείχνει ποια είναι η εμπορική προέλευση προϊόντων που διατίθεται στην αγορά. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πολλές φορές επιμείνει και υπενθυμίσει ότι αυτό είναι ο ρόλος του σήματος. Υπάρχει λοιπόν νομοθεσία για τα σήματα, νομοθεσία η οποία επιτρέπει στις ε, επιχειρήσεις να ε, προστατεύονται από ένα, διακριτικό, ένα διακριτό μάλλον σήμα ε, ένα σήμα που επιτρέπει την αναγνώριση και την προστασία τόσο του καταναλωτή όσο και του παρακοκού από τον αθέμητο ανταγωνισμό και την αθέμητη διάθεση στην αγορά. Έτσι μπορούμε να εκφράζουμε ως καταναλωτές την προτίμησή μας για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με βάση την επιλογή του σήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέξουμε τις επενδύσεις στους ε, λοιπούς τομείς, αλλά ιδιαίτερο μέλημα θα πρέπει να δώσουμε στην, για την προστασία της διαφάνειας της αγοράς. Πέραν αυτού, και με σεβασμό τη νομοθεσία που είναι ενισχύει, θα πρέπει να γίνει σεβαστή και η ελευθερία τη ενημέρωση και πληροφόρηση. Δηλαδή, εν ολίγης, δύο συμφέροντα των πολιτών που αξίζουν και τα δύο ε, προστασίας δεν πρέπει να έρθουν σε αντιπαράθεση, σύγκρουση ή να χρειαστεί να επιλεγεί το ένα έναντι του άλλου. Δηλαδή το να θέλουμε να προστατεύσουμε το σήμα δεν ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να παρεμποδίσουμε σε απόλυτο βαθμό την χρήση του σήματος από κάποιον άλλον. Απλώς πρέπει να προστατεύουμε τα προϊόντα που καλύπτει το σήμα. Επίσης, ίσω θα πρέπει να διευρύνουμε τον αριθμό των υποκειμένων δικαίου που έχουν το δικαίωμα να κάνουν ε, την ε, ένσταση προσφυγή, να αντιδράσουν δηλαδή στην ε, αντιγραφή του σήματος. Πολλές φορές μετά την δημοσίευση ενός αιτήματο μπορούν να παρέμβουν οι εμπλεκόμενοι στην αγορά για να, πούν, να εξηγήσουν λόγους του οποίου θα πρέπει να αποκλειστεί από, την, από το πεδίο εφαρμογή νομοθεσία ένα συγκεκριμένο σήμα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει ο καθένα από αυτά τα υποκείμενα δικαίου να είναι σε θέση εξ αρχή να επισημαίνει τι παρατηρήσει του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα κίνδυνο να παρασυρθεί σε μια ε, παρεξήγηση ω προ τα χαρακτηριστικά του προϊόντο και το συγκεκριμένο σήμα ο καταναλωτή. Αυτέ είναι οι παρατήρησει που είχα για την έκθεση. Παρακαλώ την εισηγήτρια να τα λάβει υπόψη. Φυσικά θα τι καταθέσω και με τη μορφή τροπολογιών. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. κύριο Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικά γενικά σχόλια, καταρχά. Εκ μέρου του κύριου Κρότσμαν. Χαιρετίζουμε τι θέσει τη εισηγητρίας και κυρίω την υποστήριξη που εκφράζει στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα που αφορούν τι αρμοδιότητε τη Επιτροπή μα και ειδικότερα την ενίσχυση των δικαιούχων στον αγώνα για, την καταπολέμηση των απομήνυσεων από τρίτα κράτη που χρησιμοποιούν ω κέντρο διακίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούν να πουλήσουν μέσα σε αυτήν τα προϊόντα του. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία για τα σήματα, μεγάλο τμήμα των προτάσεων τη κυρία Μπαστό ε, το υποστηρίζουμε, ιδιαίτερα εκεί όπου γίνεται λόγο για την υποστήριξη από τις εθνικές αρχές του δικαιούχου στη διαδίκηση των προϊόντων, των ε, συμφερόντων τους και την ε, καταχώρηση του σήματος. Δεν συμφωνούμε όμως ότι θα πρέπει οι διεθνείς ε, υπηρεσίες σήματος να εξετάζουν όχι μόνο τα απόλυτα αλλά και τα σχετικά εμπόδια στην, στην καταχώρηση. Νομίζουμε ότι αυτό θα σήμαινε η αυτεπάγγελτη δηλαδή εξέταση των σχετικών εμποδίων ή κολλημάτων καταχώρησης θα σήμαινε πολύ μεγάλο γραφειοκρατικό και οικονομικό βάρος για τις υπηρεσίες σήματος. Αυτό πρέπει να δετίθεται μόνο κατόπιν, ε, σαν υπηρεσία κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου. Α, ήρθε ο κύριος Κρόιτσμαν. Α, ας συνεχίσω ο Και περνάω τώρα στον κανονισμό για τα σήματα. Ελπίζω ότι καλύπτω όλες τις παρατηρήσεις. Χαιρετίζουμε την πρόταση της συγγήτριας ε, για την προστασία της προστατευομένης ονομασίας προελεύσεως και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών από και τη μεταφορά του ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Εναρμονισμένη Υπηρεσία για την Εσωτερική Αγορά, πράγμα το οποίο μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα στην προστασία αυτών των ονομασιών. Επίση, θέλουμε το Διοικητικό Συμβούλιο να ε, λάβει υπόψη τι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε περίπτωση σημαντικών ε, πλέον ασμάτων να περιορίζει το κόστος για την καταχώρηση αυτή. Τέτοιου είδους όμως ποσά δεν θα πρέπει να ε, εισραίουν στη συνέχεια στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να αφιερώνονται ειδικά στην προστασία της πνευματικής διοκτησίας. 96,3% των αιτήσεων για την πνευματική ιδιοκτησία έγιναν με ηλεκτρονικό τρόπο τελευταία χρονιά και είναι πολύ πιο απλή αυτή η διαδικασία. ω εκ τούτου δεν χρειάζεται πλέον να περνούν οι αιτήσει από τις εθνικές υπηρεσίες σε αυτό διαφωνούμε με την εισηγήτρια. Νομίζουμε ότι είναι πολύ πιο οικονομική η ευρωπαϊκή προσέγγιση και μας ε, επιτρέπει να δαπανούμε λιγότερα από τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Φορολογουμένου. Πιστεύουμε ότι με την νέα υπηρεσία μπορούμε να έχουμε προστασία των προϊόντων ε, με βάση και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικοστηρίου και μετά την περίοδο που ορίζει σχετική απόφαση να ισχύει το σήμα με βάση τη συγκεκριμένη ε, ταξινόμηση και ονομασία. Η εισαγωγή τροποποιήσεων που προτείνει η εισηγήτρια είναι, πιστεύουμε, ζήτημα του δικαιούχου. Και αυτό σημαίνει ότι προτιμούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν δεχόμαστε τροπολογίες. Αλλά θα πρέπει η δυνατότητα για την προσαρμογή, η διόρθωση να επεκταθεί από τους 4-12 μήνες για να έχει περισσότερο χρονικό περιθώριο στη θέση του ο δικαιούχος. Πάντως οι διαφορές που ε, εντοπίζουμε δεν είναι τεράστιες και έτσι πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Κύριε Κρότσμαν, αν έχετε τίποτα να συμπληρώσετε. Όχι, Πρόεδρε, ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη γιατί έπρεπε να πάω στην Επιτροπή Μηχανία να μιλήσω εκεί. Του είχα όμω ε, δώσει του Γιώργου το, την ομιλία μου. Κύριε Σέγκστρομ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η ουσία των εμπορικών σημάτων είναι η διευκόλυνση του νομότυπου εμπορίου και να βελτιωθεί η ευρύθμινη λειτουργία της αγοράς, της εσωτερικής αγοράς εν προκειμένου. Όμως πράγματι ο σκοπός ε, του συστήματος της ύπαρξης εμπορικού συστήματο εμπορικών σημάτων είναι αυτή η διευκόλυνση. Δυστυχώ η πρόταση τη Επιτροπή έχει δύο στοιχεία που κινούνται προ την αντίθετη κατεύθυνση. Πρώτον, θέλουμε να παρατείνουμε και να διευρύνουμε το δίκαιο εμπορικού σήματος ε, όχι μόνο δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια αλλά και στα εμπορεύματα, στα διαμετακόμιση. Αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τα, ε, τα παραποιημένα γιατί είναι ήδη παράνομο και ε, οι εγκληματίε δεν ακολουθούν ε, το νόμο, επομένω δεν έχει νόημα να πούμε ότι για άλλη μια φορά είναι παράνομη αυτή η δραστηριότητα. Όμως η επέκταση ε, του δικαίου για να καλύπτουμε λιμένε όπω το Ρότερνταμ και άλλοι, ε, Έχουμε πρώτο το ζήτημα εκεί της πρόσβασης στις φαρμακευτικές ουσίες. Ήδη είδαμε φορτία με φάρμακα προς χώρες του τρίτου κόσμου έχουν ε, κατασχεθεί λανθασμένο, ε, λανθασμένα εξαιτία ε, του δικαίου εμπορικών σημάτων και αυτό θα μεγεθύνει τέτοιου είδου προβλήματα. Τα τελωνία στο Ρότερνταμ και αλλού θα έχουν περισσότερα εμπορεύματα να ελέγξουν στο νόμιμο εμπόριο και αυτό δεν έχει νόημα γιατί όταν πάμε σε τρίτη χώρα όπου δεν υπάρχει εμπορικό σήμα, τότε δεν υπάρχει λόγος να κατασχεθεί στη διαδικασία της διαμετακόμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς και μόνο επειδή δεν έχει εμπορικό σήμα. Νομίζω ότι αυτό θα βλάψει το νόμιμο εμπόριο και νομότυπο εμπόριο στην Ευρώπη. Και δεύτερον και ακόμα χειρότερο, είναι η πρόταση και πάλι επέκταση ε, των δικαιωμάτων ε, των τελωνικών αρχών και των καθηκόντων των τελωνικών αρχών για κατάσχεση δίμευση προϊόντων που έχουν ε, αγοράσει μεμονωμένοι αγοραστές στο διαδίκτυο. Εάν εγώ ως αγοραστής αγοράσω κάτι από ένα site στο Χονγκ Κονγκ στην Αμερική, δεν έχει σημασία ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό απολύτως ε, νομότυπο, κατασκευασμένο από την εταιρεία, αλλά εγώ το αγοράσω εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε βάσει τη υφιστάμενη αυτής πρότασης, τα τελωνία θα πρέπει να κατασχέσουν το προϊόν. Αν ε, εγκριθεί αυτή η πρόταση, ο μέσος καταναλωτής δεν γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ των ξένων site εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ρωτήσετε κάποιο στον δρόμο, κανένας δεν θα γνωρίζει με σιγουριά που έχει την έδρα της η Amazon, για παράδειγμα, αν είναι εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές θα αγοράζουν νομότυπα ε, προϊόντα, θα ε, κατάσχονται από τα τελωνία και θα πούν σε όλους ε, τους ε, φίλους τους, στον κύκλο τους, ότι δεν πρέπει να, δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι το εμπόριο στο διαδίκτυο γιατί τα τελωνία θα στο κατασχέσουν. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και όπως έχει αναφερθεί και πολλές φορές στην Επιτροπή μας, πώς θέλουμε να προαγάγουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιο. Τώρα, άλλα σχόλια ίσονος σημασίας, γιατί τα πρώτα δύο τα θεωρώ εξαιρετικά σημαντικά. Ναι, συμφωνώ με τον κύριο Πανσέρη για την ελευθερία έκφρασης. Αυτή τη στιγμή, στο ουσιώδες ε, δίκαιο εμπορικών σημάτων, αν εγώ, ας πούμε, θέλω να χρησιμοποιήσω ένα εμπορικό σήμα σε πολιτιστικό έργο ή για σκοπούς ψυχαγωγίας, έχω το δικαίωμα να το πράξω. Όμως, υπάρχει μεγάλη κατάχρηση όταν οι δικηγόροι εμπορικών σημάτων εσφαλμένα ισχυρίζονται ότι δεν μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Το τελευταίο παράδειγμα ήταν πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία. Υπήρχε μια αντίστοιχη ε, αφίσα που έχει γίνει πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, παρότι χρησιμοποιήθηκε και αρχικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, κάποιος λοιπόν έχει βρει αυτή την αφίσα και απειλεί όσους θέλουν να αναπαράξουν αυτή την αφίσα ή όσους θέλουν να το τυπώσουν σε μπλούζες και το καθεξής ότι αυτό αντιβαίνει στο δίκαιο εμπορικών σημάτων. Αυτό δεν έχει καμία νομική βάση. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν αυτό. Επομένω, αν κάποιο λάβει μια απειλή από έναν δικηγόρο εμπορικών σημάτων που προσπαθεί να καταχαραστεί του δικαίου, οι περισσότεροι απλώ ε, παρετούνται και επαναχωρούν. Συμφωνώ λοιπόν με τον κ. Πανσέρη ότι θα ήταν πολύ χρήσιμη μια διευκρίνηση ε, για να τονίσουμε ότι το εμπορικό σήμα ε, περιορίζει μόνο την χρήση εμπορικού σήματος. Δηλαδή όταν κάποιος χρησιμοποιεί ένα σήμα που ταυτοποιεί ένα προϊόν που βρίσκεται στην αγορά. Αυτή η διευκρίνηση θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Συμφωνώ ε, και με την εισηγήτρια για την οδηγία εμπορικών σωμάτων, γιατί η Επιτροπή θέλει να απαγορεύσει τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, έρευνα εξ Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Πρώτον, προσωπικά θεωρώ ότι οι έρευνε εξ εντάξει, υπάρχουν ε, επιχειρήματα υπέρ και κατά. Εγώ τίνω ε, να θεωρήσω ότι είναι κάτι το ωφέλιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως και πάλι υπάρχουν και επιχειρήματα κατά. Όμως αυτό θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Υπάρχουν ε, διαφορετικά ζητήματα στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιβάλλουμε μια ενιαία λύση σε όλα τα κράτη-μέλη από τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, να διαφωνήσω με την ε, εισηγήτρια σε ό,τι αφορά ε, τις χρεώσεις. Ε, νομίζω ότι το πλεόνασμα θα πρέπει να επιστρέφει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας οργανισμός όπως όλοι οι υπόλοιποι. Οι υπεστήριοι οργανισμοί χρειάζονται χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, του τα δίνουμε. Αυτό ο οργανισμό έχει ένα πλεόνασμα και πιθανότητα να συνεχίσει να έχει πλεόνασμα και στο μέλλον. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λογικό είναι για μένα. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι με, αυτές τις, με αυτά τα τέλη πρέπει να τα ε, μειώνουμε να δυνατόν ε, περισσότερο για να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν ισχύει για τα εμπορικά σήματα όμως. Στα τέλη εφαρμογή βεβαίω θέλουμε να τα, να τα κρατήσουμε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, όμως θα πρέπει να καλύπτεται το κόστος της αίτηση. Όμως για τα τέλη ανανέωση δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα φτηνά και χαμηλά. Γιατί στην ανανέωση έχουμε ένα εμπορικό σήμα για 10 χρόνια, μετά ξέρει κάποιο αν πρόκειται για επιτυχέ σήμα ή όχι. Ιδάλω δεν πρόκειται να το ανανεώσει κανεί. Αν είναι επιτυχέ. Προφανώ ε, όποιο τα έχει εδώ για 10 χρόνια θα έχει ε, βγάλει αρκετά χρήματα για να πληρώσει και μερικέ εκατοντάδε ευρώ δεν θέλουμε να είναι πολύ χαμηλά, γιατί τότε ε, θα υπάρχει μια ανανέωση έτσι κι αλλιώς. Και θα παραμείνουν πολλά εμπόδια στα μητρό εμπορικών σημάτων που ε, δεν βοηθά κάποιες επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν εμπορικό σήμα. Λοιπόν, για τα τέλη. θα θέλουμε να ε, έχουμε τέλη που να συνεχίσουν να δημιουργούν πλεόνασμα, το οποίο είναι βεβαίω πολύ καλό να υπάρχει και για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Oh, thank you for some very pertinent... Σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ εύστοχα τα σχόλιά σας. Ο κύριο Μπιέλαν τώρα, ο τελευταίο μα και ο Και μετά ποιος άλλο επιθυμεί το λόγο από τα μέλη τη επιτροπή ευπρόσδεκτο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια των γνωμοδοτήσεων. Των γνωμοδοτήσεων που αφορούν την οδηγία και τον κανονισμό. Έχουμε ελάχιστο χρόνο, σύντομε λοιπόν παρατηρήσει. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις τροπολογίες ε, της συγγήτριας. Χαίρομαι που προσπαθεί η συγγήτρια να τροποποιήσει το άρθρο 41 για τις αυτεπάγγελτες ε, έρευνες. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να διαγραφεί ολόκληρο το άρθρο. Εγώ θα προτιμούσα το θέμα αυτό να το αφήσουμε στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να θα κάνουν τέτοιε αυτεπάγγελτε έρευνε και θα υποβάλω και σχετική τροπολογία. Έχω κάποιε επιφυλάξει και για την οδηγία και για τον κανονισμό. Για παράδειγμα, το άρθρο, τα άρθρα 52 και 53 της οδηγίας ε, που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών οργανισμών και του κοινοτικού οργανισμού. Δεν το ανέφερε αυτό η συγκεντρία. Εγώ είμαι υπέρ τη στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αργών και του κοινοτικού οργανισμού και μάλιστα το ανέφερε και στην γνωμοδότησή μου για το παρατηρητήριο. Αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να κρατήσουμε κάποια ελαστικότητα, να αφήσουμε κάποια ευελιξία στι εθνικέ αρχέ για το πώ θα δώσουν σάρκα και οστά σε αυτή τη συνεργασία με το κοινοτικό οργανισμό. Και για το σημείο αυτό λοιπόν θα υποβάλω τροπολογίε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό. Έχω διαφορετική γνώμη για το άρθρο 123 γάμα, 2, 3 και 4 εδάφια που αφορά τις ε, ε, επιχορηγήσεις και δεν ξέρω πόσες, ε, ε εθνικά γραφεία ή ε, πόσο μπορούν να επηρεάσουν το κοινοτικό πρόγραμμα γιατί και πάλι για τα κονδύλια ε, και τα τέλη, δεν ξέρω, θα πρέπει να τα κρατήσουμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για τις κατεξουδιώτες πράξεις, ε, θα ήθελα κάτι τέτοιο να μπει στον ίδιο τον κανονισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, οργάνωση, έχει υποβάλει η συγγήτρια μια τροπολογία για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, συμφωνώ και επίσης για το θέμα διορισμού και ανάκλησης ε, του εκτελεστικού διευθυντή. Το σχέδιο κανονισμού λέει ότι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να λάβει την απόφαση για την ανάκληση του εκτελεστικού διευθυντή. Εγώ δεν συμφωνώ με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποβολή της αίτησης ε, και θα υποβάλω και σχετική τροπολογία. Σας ευχαριστώ. Oh, Ευχαριστώ πολύ. Τους ο θέλει κανείς άλλος να κάνει σχόλια. Ίσως αν με ακούσει ο κύριος Κρόιτσμαν και να μην ε, συνομιλεί με τον κύριο Χατζημαρκάκη. Νομίζω ότι θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να ακούσουμε τα σχόλια του κυρίου Έγκστρομ για την ε, σχέση μεταξύ της δικής σας προτάσεως και της ε, άλλης προτάσεως για το θέμα της πνευματικής διοκτησία και του ε, αντιμετώπιση μετακόμισης και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρηση του κυρίου Έγκστρομ ότι οι ορισμοί γιατί πού μπορούν οι τελωνιακές αρχές να παρεμβαίνουν για την προστασία της πνευματικής διοκτησία είναι ε, απαραίτητο να ενσωματωθούν εδώ. Και επίση η αρχική πρόταση της Επιτροπής ε, ότι μπορούν οι τελωνιακές αρχέ να παρεμβαίνουν για να ε, παρεμποδίζουν τη διακίνηση προϊόντων και σημάτων που βρίσκονται πριν από την εκπνοή και μέσα και έξω στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε αυτό και να το ενσωματώσουμε. Εμένα με απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα τη εκπνοή του σήματος. Γιατί αποτελεί βέβαια περιορισμό, όπω είπε ο κ. Σέγγστρομ, τη ελευθερία του ιδιώτη για τον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν θα σας παρακαλέσω για ένα σχόλιο. Λίγα λεπτά μας έχουν μείνει ακόμα. Παρακαλώ τον κύριο Κιόνιχ να λάβει το λόγο. Γρήγορα όμως και σύντομα, γιατί το άλλως θα τα ξαναπούμε με τις τροπολογίες. Και μετά θα δώσω το λόγο και στην κυρία Μπάστος. Κύριε Κιόνιγκ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ. Δεν είμαι ο κύριος Κιόνιγκ ωστόσο. Είμαι ο Τόμας Άχινμπεργκ από την ε, μονάδα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Γενικής Δεύθυνσης για την Ιστορική Αγορά. Σύντομος θα είμαι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τη γενική υποστήριξη που εκφράζει για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο συγκητής. Στόχος είναι να ενισχυθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη και να γίνει η Ευρώπη μια πιο ανοιχτή, αποτελεσματική και δεκτική αγορά και ασφαλής αγορά για τις επιχειρήσεις. Χρειάζεται μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση των προϊόντων αναπομίμησης, κυρίως κατά τη μεταφορά και τη μετακόμιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει εν προκειμένου ότι πρέπει να αποφύγουμε την μετατροπή της Ευρώπης σε ένα ε, κόμβο από τον οποίο θα διέρχονται τα προϊόντα απομίμησης για να μεταφερθούν στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αλλά όχι με το σήμα, με την ομοθεσία για το σήμα. Υπάρχει περιδιοφόρο για περαιτέρω βελτίωση και ανάγκη για πιο ακριβή διατύπωση στο θέμα της ε, δράσης ή παρέμβαση των τελωνιακών αρχών, πολύ φορές να το κοιτάξουμε. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε τις ε, προσπάθειες των εισηγητών και θα θέλαμε να ε, προχωρήσει και να βελτιωθεί ασφαλώς όλη αυτή η δέσμη μέτρων. Υπάρχουν μέτρα για τις βιομηχανικές για τις πτυχές βιομηχανικής και, και οικονομικής πολιτικής που θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά και αν μου επιτρέπετε Πρόεδρε ένα-δύο σημεία πιο συγκεκριμένα να θίξω. Μας έχουν απασχολήσει και στη σχέση με ορισμένους ομιλητές. Καταρχάς, για τους εισηγητές η επιλογή της ε, ε, αίτηση για προστασία σήματος ε, για, τον, ε, η κατεπιλογή δηλαδή υποβολή της αίτησης είναι κάτι το οποίο δεν αποσκοπεί τόσο να διευκολύνει τη δουλειά, τη, τη, ζωή του επιχειρηματία, όσο στο να γίνει σωστά η δουλειά. Οι περισσότερε αιτήσει αυτή τη στιγμή, το 96% και 100 των αιτήσεων για το 2012, έχουν περάσει από το ηλεκτρονικό σύστημα, ωστόσο. και να εξετάσουμε και ποια είναι η λογική που διέπει αυτόν τον κανονισμό. Το καθεστώς της έγγραφης αίτησης ήταν μεταβατικό. Είχε στόχο να ε, βοηθήσει τον ε, ετούντα σε μια περίοδο που δεν ήταν γνωστό το κεντρικό, δεν ήταν γνωστή η κεντρική υπηρεσία και θα τον ε, απαλλάσαμε από περιττές μετακινήσεις ενδεχομένω και ταλαιπωρία. Τώρα όμως μπορεί να γίνει μέσω της, ε, του, δικτύου αυτή η αίτηση και θα πρέπει να διευκολυνθεί περισσότερο αυτή η διαδικασία παράγραπτη. η ευελιξία ως προς την καταχώρηση από τους διαφόρους δικαιούχους νέων υπηρεσιών ε, ή δυνατοτήτων που ζητήθηκε. Θα θέλαμε να πούμε ότι θα πρέπει να επιτρέψει στο ταχύτερο, το, ταχύτερο δυνατό σε όλους τους εμπλεκομένους και δικαιούχους να προσαρμόζουν τις προτάσεις τους. Σε σχέση με την οδηγία για την προστασία του σήματος, του εμπορικού σήματος, οι παρατηρήσεις μου είναι οι εξής και κυρίως μία πολύ σημαντική πρόταση για μία κοινή προσέγγιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με μία αυτεπάγγελτη εκτίμηση για, μένα θα πρέπει, για μας θα πρέπει να καταργηθεί. Η προσέγγιση μας ήταν ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλιστεί ένα κοινό πεδίο ανταγωνισμού και εναρμόνιση για τα υφιστάμενα συστήματα σήματος. Το να δημιουργηθούν νέα ή επιπλέον υποχρεώσεις και πάνω απ' όλα διαφορετικές προσεγγίσεις στην καταχώρηση νέων σημάτων που θα οδηγούσαν και σε προσφυγές και σε ενστάσεις ε, δεν είναι καλή λύση. Η εξέταση των σχετικών χαρακτηριστικών ε, θα πρέπει να προκύπτει κατόπιν ετήσεω του ενδιαφερομένου και όχι αυτεπάγγελτα. Αυτό που μας ενδιαφέρει, θέλουμε να, υπογράψουμε, να υπογραμμίσουμε βέβαια, είναι όχι να εκθέσουμε σε ενδεχόμενες επιθέσεις ή κινδύνους του δικαιούχου, αλλά να επιτρέψουμε στις ε, αρμόδιες υπηρεσίες να ε, διερευνούν αυτές τις επιπτώσεις ε, ή τα έμεσα χαρακτηριστικά μόνο κατόπιν ετήσεω, ώστε να μην έχουν υπερβολική επιβάρυνση. Επίσης, η υπηρεσία θα πρέπει και στο μέλλον να αναλάβει και την καταχώρηση γεωγραφικών προελεύσεων που αυτή τη στιγμή έχει στις αρμοδιότητες ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία πρόταση η οποία μας φαίνεται ενδιαφέρουσα, δεν θα ήταν κακό να την μελετήσουμε, αλλά πάλι δεν θέλουμε να ε, επιβάλλουμε υποχρεωτικό γραφειοκρατικό φόρτο σε όλη αυτή την ε, προσπάθεια. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προτάσεις του εισηγητού στο θέμα αυτό ενδέχεται να ε, σημάνουν αρκετά σημαντική επιβάρυνση. Εμείς θέλαμε αυτό το νομοθέτημα, αυτή τη δέσμη προτάσεων να παραμείνει ισχνή σχετικά και να προχωρήσει στην ικανοποιητική προστασία από την απομίμηση των σημάτων της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Σεγέτηρα, δυστυχώς έχει εξαντληθεί ο χρόνος. Ε, δεν προλαβαίνετε να κάνετε τη σύνοψη. Εκτός αν ε, σε ένα λεπτό μπορείτε να κάνετε μια πολύ σύντομη ανακεφαλαίωση στον πιο βασικό σημείο. Γιατί ήδη μας παραχώρησαν ε, επιπλέον λεπτά οι διερμηνείς, αν και κάναμε προηγουμένω ε, δύο διαλύματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ λακωνική να ευχαριστήσω θερμά του συναδέρφους ε, για τις ε, προτάσεις του και τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τι διευκρινήσει του. Θα ήθελα να συνοψίσω σε δύο λόγια τις ανησυχίε μου για το κεντρικό θέμα που ενδιαφέρει την Επιτροπή μας και το μήνυμα που θα πρέπει να στείλουμε προς τους ε, συμπολίτες μας. Με την αναθεώρηση αυτή των δύο νομοθετικών κειμένων θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην αγορά. Να μην συνεχίσει η Ευρώπη να είναι παράδεισος, να είναι παράδεισος για την πειρατεία, την απομίμηση και την παραποίηση και να κάνουμε πιο ευέλικτα τα θεσμικά συστήματα εμπορικού συστήματος, ώστε και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα με πιο εύκολο και μη δαπανηρό τρόπο. Για ορισμένα σημεία και τροπολογίε θα είμαι ιδιαίτερα ε, διαλλακτική, αλλά σε άλλα όχι τόσο. Το θέμα των αγαθών σε διαμετακόμιση είναι πολύ εύστοχο. Επίσης το θέμα των ε, αγορών μέσω διαδικτύου. Εδώ έχουμε διάσταση απόψεων ε, και διαφορετικές ε, γνώσεις, ε, απόψεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δώσουμε τα σωστά μηνύματα και στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά όλους και ιδιαίτερα την εισηγητριά μας για να σα υπενθυμίσω την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών που λέγει αύριο 26 του μηνό στι 12 το μεσημέρι. Η εξέταση των τροπολογιών θα γίνει στι 14 Οκτωβρίου και θα ψηφίσουμε στι 5 Νοεμβρίου. Ενώ στι 26 θα ψηφίσει η αρμόδια καθήλια επιτροπή, νομική επιτροπή. Ραντεβού στι 3 η ώρα με, πρόεδρο την κυρία Πιετικάινεν, την οποία ε, ευχαριστώ και σας ε, παρατρύνω να είστε στην ώρα σα όλε τι 3. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.